τον συντάξαντα, τον κύριο Κώστα, για πέντε λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ, παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, η Επιτροπή της οποίας εσείς είστε μέλος επανειλημμένως ανακοίνωσε το πρόγραμμά της για την αστική κινητικότητα και το οποίο θα έπρεπε να υποβληθεί από τον περασμένο φθινόπωρο στην ε, Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η Κομισιόν ανέλαβε αυτή την ευθύνη και ολοκλήρωσε τη διαβούλευση για το πράσινο βιβλίο για την ε, αστική κινητικότητα που ξεκίνησε το 2007. Το επανέλαβε στο πρόγραμμα δράσης για ε, τις υποδομές για τις μεταφορές εμπορευμάτων. Το επανα... Το επανέλαβε για τον εσωτερήκευση του εξωτερικού κόστους για τις μεταφορές του 2008 σε σχετικό πλάνο, αλλά ο χρόνος κυλά και δεν βλέπουμε το πρόγραμμά σας. Εμείς φοβούμαστε με το τέλος της θητείας ότι πολλή από τη δουλειά που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια θα απεβεί εις Κυρία Επίτροπε, μπορείτε να με διαβεβαιώσετε, μπορείτε να μου πείτε πώς θα δημοσιοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες ώστε να μπορέσει τούτο εδώ, τούτο εδώ το σώμα να οριστικοποιήσει τις συστάσεις του αυτές που περιλαμβάνονται στο ψήφισμα ΡΑΚ για μια νέα κουλτούρα αστικής κινητικότητας που ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2008. Κυρία Επίτροπε, η αστική κινητικότητα είναι αναμφίβολα ένα φαινόμενο το οποίο εμφανίζεται τοπικά και το οποίο πάντοτε θα βλέπει την τοπική αρμοδιότητα να κυριαρχεί της εθνικής και της κοινοτικής της ε, Ευρωπαϊκής. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει καμία κοινοτική ή κρατική παρέμβαση και ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα ε, μπορεί, θα οφείλει να ορίσει το ρόλο της ίδιας σε αυτό το πλαίσιο η αδράνεια της Κομισιόν δεν βοηθά στις μεταφορές, στις αστικές μεταφορές, ούτε στην αντιμετώπιση της ρήπανσης της πόλης και ξέρουμε ότι πάνω από το 40% των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα προέρχονται από τις αστικές μεταφορές ε, και ότι έτσι δεν βοηθάμε ούτε την ασφάλεια στους δρόμους. Πολλά από τα θανατηφόρα ατυχήματα ε, προκαλούνται στις πόλεις. Ούτε προστατεύονται οι καταναλωτές, οι πιο αδύναμοι ε, πολίτες, οι οποίοι, των οποίων η κινητικότητα εξαρτάται εξαρτάται από τις αστικές μεταφορές. Μπορούμε να περιμένουμε από το κράτος μέλος, από το ένα κράτος μέλος στο άλλο κράτος μέλος, από τη μία πόλη στην άλλη. Κυρία μου, σε εσά απευθύνομαι. Από τη μία πόλη στην άλλη για την επεράσπιση του αστικού περιβάλλοντος, να επιμείνουμε για την προστασία της κινητικότητας των πολιτών. Μήπως είναι αυτά τα δικαιώματα τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συμβάλλει ώστε να τα εγγυάται σε όλους τους Ευρωπαίους. Δηλαδή, προδιαγραφές, στόχοι, ομοιόμορφοι, σωστές πρακτικές, συντονισμός των μέσων, η εκπόνηση αξιόπιστων στατιστικών δεν είναι αυτός ένας χώρος που αν τον ανακαλύψει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βοηθήσει την επικουρικότητα για τα οποία, ε, την οποία τα κράτη-μέλη και οι τοπικές αρχές έχουν κάθε δικαίωμα να είναι περήφανα. Τώρα, ε, θα πρέπει να μας εξηγήσετε τους λόγους της καθυστέρησης ε, που αγγίζει τα όρια της αμέλειας για την αστική κινητικότητα. Θα πρέπει να μας πείτε γιατί δεν τηρήσατε αυτήν την ε, υπόσχεσή σας. Πρόκειται για πραγματικά για αιτίες ή για ευθυνές δικαιολογίες. Η Κομισιόν μήπως έχει γίνει τόσο συνετή που τελικά αρνείται να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των ευρωπαϊκών λαών ε, για να μην ενοχλήσει τα κράτη. Αυτοκτονική μου φαίνεται αυτή η στρατηγική. Μετά από το εξαιρετικό εξάμεινο της Γαλλικής ε, Προεδρίας που ήταν ένα φωτεινό παράδειγμα. Όλο για delivery και contra delivery μας μιλάτε. Δηλαδή απόδοση και παραγωγικότητα. Το μικρό παράδειγμα αυτού του προγράμματος για την αστική και γεννητικότητα μπορεί να δώσει ένα παράδειγμα για την επίλυση αυτού του ευρύτερου προβλήματος. Σας ευχαριστώ. Ε, κύριε Βασιλείου, για το λόγο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα-πρώτα Θέλω να σας πω ότι ο Αντιπρόεδρος Ταγιάννη ζητεί συγγνώμη που δεν μπόρεσε να παραστεί στη συζήτηση διότι είχε μια πάρα πολύ σημαντική αποστολή να επιτελέσει στην Ιαπωνία και τώρα επί τη ουσία του ζητήματο, πρέπει να σα πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 100% έχει δεσμευθεί να συνεχίσει την πολιτική που χαράξαμε όσον αφορά την κινητικότητα διότι είμαι θα πεπισμένη ότι παρά το ότι ε, η βασική αρμοδιότητα την έχουν οι τοπικές, οι περιφερειακές και εθνικές αρχές. Για κάποια συγκεκριμένα ζητήματα υπάρχει προστιθέμενη αξία όσον αφορά την ανάληψη δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ε, παρά το ότι κάθε πόλη έχει τις δικές της ε, ιδιορυθμίες, όλοι έχουν τις κοινές προκλήσεις ε, η κινητικότητα είναι κάτι το οποίο συνέχεια γίνεται πιο σημαντικό, αφορά όλο τον κόσμο, έχουμε τα προβλήματα τα συγκοινωνιακά, έχουμε την προσβασιμότητα στην δημόσια συγκοινωνία, έχουμε ε, την, την, την μόλυνση της ατμόσφαιρας και για να καταλάβετε πόσο σημαντική είναι η κινητικότητα να σας πω κάποια στοιχεία. Έχουμε 60% του πληθυσμού που μένει σε αστικό περιβάλλον στις πόλεις, το 85% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί ε, παράγεται. Όμως οι πόλεις ευθύνουν για το 40% των εκπομπών του διοξιδίου και δύο από τα τρία τροχέα συμβαίνουν σε αστικές περιοχές. Τέλος, ε, αυτή η κυκλοφορική συμφόρηση είναι βασικό πρόβλημα που το αντιμετωπίζουν οι κάθε μέρα. Και η συμφόρηση οφείλεται συγγνώμη, ευθύνεται για την απώλεια 100% του ΕΠ. Οπότε χρειάζεται μια βιώσιμη κινητικότητα, κατά το οποίο είναι το κλειδί για να πετύχουμε του στόχου μα όσον αφορά τι αλλαγέ ε, του κλίματο, τη οικονομική ανάπτυξη και τη ε, αγωτική ασφάλεια. Οπότε και εμεί έχουμε χαράξει κάποιο πρόγραμμα δράσεων από το 1995 και έτσι θέλουμε να έχουμε ανταλλαγή των αρίστων πρακτικών. Και έχουμε το πολύ αξιόλογο πρόγραμμα Civitas, το οποίο το 2000, το 2007 ε, έχουμε μια πράσινη βίβλο η οποία ε, χαράξει καινούργιο δρόμο στην κινητικότητα και γι' αυτόν τον τρόπο έχουμε κάποιες συμπληρωματικές δράσεις σε ενωσιακό επίπεδο ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ε, πόλεις πιο φιλικές στο περιβάλλον και επίσης να είναι δημόσιες κοινωνίες πιο εύκολα προσβάσιμες. Να δούμε όμως τι μπορεί να γίνει συγκεκριμένα σε ενωσιακό επίπεδο Μπορούμε να βοηθήσουμε τις ε, τοπικές αρχές να υλοποιήσουν τις πολιτικές μας, να χρησιμοποιήσουμε όσο γίνεται καλύτερα τους πόρους της Ένωσης. Η νομοθεσία, οι καινοτόμες προσεγγίσεις και αυτές θα πρέπει να βοηθήσουν τις τοπικές αρχές ούτως ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα να βοηθήσουμε τις αγορές για τις νέες τεχνολογίες και επίσης ε, να έχουμε πιο περιβαλλοντικά αυτοκίνητα, πιο πράσινα αυτοκίνητα, να έχουμε καλύτερα πρότυπα όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες που θα πρέπει να μπουν σε, στην αγορά. Επίσης, θα πρέπει να βοηθήσουμε τις τοπικές αρχές για κάποιες διαλειτουργικές λύσεις και να διευκολύνουμε την πιο εύρεθμη λειτουργία της ενιαίας αγορά Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειές της, διότι πιστεύει, όπως και περισσότερο από τους εμπλεκομένους, ότι πολλά πρόκειται να κερδίσουμε εάν σε ενωσιακό επίπεδο προσπαθούμε και έτσι ε, σε κάθε επίπεδο αναλάβουμε πρωτοβουλία. Τώρα να σας απαντήσω αυτό το οποίο ρωτήσατε γιατί. Αργήσαμε να λάβουμε την πρωτοβουλία. Αυτό έγινε διότι δυστυχώς δεν υπήρχαν οι κατάλληλες ε, συνθήκες ώστε να έχουμε ένα πρόγραμμα δράση ολοκληρωμένο μέχρι ότου φτάσουμε στο τέλος του 2008. Όμως ο Αντιπρόεδρος και συνάδελφος Ταγιάννη σας διαβεβαιώνει ότι είναι πάγια δέσμευσή του όσον αφορά αυτό το πρόγραμμα δράσης και όσον αφορά το να υπάρχει ε, ένα πρόγραμμα για τις ε, μεταφορές της πόλης σύμφωνα με την αναλογικότητα αλλά και την πικρικότητα διότι δεν ε, προτιθέμεθα να έχουμε μία λύση για τα πάντα. Αντίθετα, θέλουμε να υπάρχει ένα ολόκληρο πλουστάσιο με διαφορετικά μέσα με διαφορετικά όπλα που θα έχουμε διαθέσιμο, τόσο ώστε να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα τη ερδημίες κάθε πόλη και να λύσουμε το πρόβλημα τη κινητικότητα. αλλά τελικά οι τοπικέ αρχέ θα αποφασίσουν τι είναι πιο δόκιμο για του δικού του στόχου για τι δικέ του ανάγκε. και για να μπορέσουμε να καλύψουμε τι ανησυχίε που ακόμα μπορεί να υπάρχουν σαν αφορά το στρατηγικό μα ρόλο για την κινητικότητα ο Αντιπρόεδρος Ταγιάννη προτίθεται να προχωρήσει σε συγκεκριμένες δράσεις ούτως ώστε να έχουμε κινητικότητα καλύτερη περισσότερη στην ε, Ευρώπη σε συνέχεια της πράσινης βίβλου, σε συνέχεια διαβουλεύσεων με τους εμπλεκόμενους οπότε και αποφασίστηκαν συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες πρόκειται να υλοποιηθούν φέτος καινοτόμε λύσεις, νέες τεχνολογίες ήδη έχει ανοίξει διαγωνισμός ε, λίγοι τέλος ε, Μαρτίου αυτή η πρόσκληση οπότε κατά 50% θα έχουμε κάλυψη των προγραμμάτων τα οποία θα είναι πιο επιλέξιμα και μόλις η σχετική οδηγία τεθεί σε ισχύ το οποίο θα γίνει περίπου τον Μάρτιο τότε θα αρχίσει ε, να λειτουργεί ένα συστότοπος όπου θα ξεκινήσουμε την πρωτοβουλία μας για πιο πράσινα οχήματα. Πληροφορία, πληροφόρηση, θα υπάρξουν και πόροι που θα διατεθούν και ανταλλαγή των αρίστων πρακτικών και έτσι θα καλύψουμε όλους τους εμπλεκόμενους αλλά και έτσι θα πιάσει τόπο το πρόγραμμα ΣΥΒΙΤΑΣ αλλά και οι σχετικές δράσεις. Επίσης, θα καταλάβουμε περισσότερο το τι, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σε κάποιες βιώσιμες πολιτικές, θα έχουμε κάποιες πράσινες ε, ζώνες και επίσης θα μπορούσαν να μελετηθούν τι ευκαιρίες υπάρχουν τόσο ώστε οι δημόσιες ε, μεταφορές να είναι πιο διαλειτουργικές επίσης. Θέλουμε να υπάρχει ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων τόσο ώστε να μπορούμε να μελετήσουμε τα διάφορα προβλήματα ε, που αφορούν το, το δικό δίκτυο και πώς θα εξωτερικεύσουν τις εσωτερικές δαπάνες και νομίζω ότι με όλε αυτέ τις πρωτοβουλίε σύντομα ε, πρόκειται να προχωρήσουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι θα αποκτήσουμε ένα θεμέλιο, μια βάση για να προοδεύσουμε όσον αφορά την κινητικότητα στις πόλεις. Η Πρόεδρος και τώρα. Να ακούσουμε τις αγορητέ των πολιτικών ομάδων και ξεκινάμε με το Ευρωπαϊκό Λοϊκό Κόμμα Ευρωπαίου Δημοκράτε. Ο κύριο Ράκ, δύο λεπτά. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επιτροπέ, με όλο το σεβασμό τη Κομισιόν γενικά και εσά προσωπικά δεν απαντήσατε πραγματικά την ερώτηση του Πρόεδρου κ. Κώστα. Μας περάσατε ένα καλό μήνυμα. Καταρχήν αναφέρατε κάτι που αναφέρεται ήδη στην Πράσινη Βίλα για την αστική κινητικότητα ότι δηλαδή χρειαζόμαστε κοινέ ευρωπαϊκές λύσεις για ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές πόλεις για οποιαδήποτε μορφή. Διαφορετικά ή με πολύ παρόμοιο τρόπο. Αυτό το είχαμε χαιρετήσει ήδη τότε, πριν από μερικούς ε, μήνες. Και οι προτάσεις Κομισιόν που μας είχαν υποσχεθεί, τις περιμέναμε με μεγάλη χαρά. Δεν έφτασαν όμως ακόμα στα χέρια μας. <coughs> Και το μόνο μήνυμα που άκουσα από εσά ήταν ότι δεν θα υπάρχει συνολικό πρόγραμμα δράσης. Τελεία. Γιατί όχι. Εάν αυτά που ακούμε και ακούμε πολλά εδώ στο σώμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό ίσως σχετίζεται με το γεγονό ότι υπάρχει ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη που ε, υποκρινόμενοι ότι εδώ υπάρχει η περισσοτερα κρατη μελη που υποκρινομενοι οτι εδω υπαρχει παρεμβαση στην επικορικότητα φοβίζουν και την ίδια την Κομισιόν φοβίζουν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις προτάσεις του είπε ρητά ότι εμείς δεν θέλουμε να παρεύουμε στην επικουρικότητα. Είπατε εσείς ότι δεν θέλετε ένα σχέδιο για όλους. Αλλά το να μην παρουσιάσουμε κανένα σχέδιο δεν είναι λύση. Και ας προχωρήσουμε λοιπόν. Ας ε, πληρώστε τις υποσχέσεις σας δεν θα εξασφαλίσετε την υπερεκλογή της Κομισιόν με το να μην γίνει τίποτα, με το να μην προσβάλλετε κάποιο κράτος, θα επανεκλεγείτε μόνο όταν έχετε υποβάλει καλές λύσεις και καλές προτάσεις. σωστική ομάδα, ο κύριος Σαβαρή, δύο λεπτά. Oui, Madame la Commissaire. Μάλιστα, κύριε Πέτροπε μόλις μας επιβεβαιώσατε και μας καθησυχάσατε στην πρωτοβουλία που συμπεριλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτό το θέμα. Μόλις είπατε ότι για προφανείς λόγους, δηλαδή λόγω της σημασίας του ότι αντιπροσωπεύουν οι αστικές μεταφορές στις μεταφορές και τους στόχους για το κλίμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να μείνει αδιάφορη για τις αστικές μεταφορές είχε αναλάβει την πρωτοβουλία με το πράσινο βιβλίο και μας υποσχέθηκε πρόγραμμα δράσης. Σήμερα δεν μπορείτε να μας το αρνηθείτε αυτό και να μας λέτε ότι το εφαρμόζεται στο πιτς φετήλι χωρίς διαβούλευση με το κοινοβούλιο, χωρίς καμιά ορατότητα ε, και καμιά διαφάνεια. Γι' αυτό το λόγο επέτυχα από τους συναδέλφους και ε, ιδιαίτερα από τον Ράιμερ Ράκ, ο οποίος καθάρισε το έδαφος, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά στη διαδικασία έχει φτιάξει το πρόγραμμα δράση που εσεί δεν θέλετε να φτιάξετε πριν από τι εκλογέ. Αυτή η πρωτοβουλία που είναι πολύ ανορθόδοξη θα έχει πολύ σημαντικό πολιτικό αντίκτυπο γιατί θα ε, ε, έρθει και θα ρωτήσει από την, στην Επιτροπή Μεταφορών το νέο επεύθυνο επίτροπο για τι μεταφορέ και θα βαρύνει πάρα πολύ στην κρίση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να θα, που σήμερα η Ευρωπαϊκή Κομισιόν υποχωρεί στην ε, ελάχιστη αντίρρηση του ελάχιστου κράτους μέλους. Και πραγματικά υπάρχει μια θεσμική ε, ε, έλλειψη. έχετε αποφασίσει να παίξετε το χαρτί της διακυβερνητικότητας και εμείς είμαστε αναγκασμένοι να διαπραγματευτούμε μεταξύ μας ένα πρόγραμμα δράσης, σας το προτείνουμε και να επιμείνουμε στο επόμενο Επίτροπος Μεταφορών να δεσμευτεί για τη συνέχεια που θα δώσει σε αυτό το πρόγραμμα δράσης. Συμμαχία των Δημοκρατών για την Ευρώπη, 2,5 λεπτά. Ο κύριος Μπουπούη, κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, με όλο το σεβασμό κύριε Επίτροπε που οφείλουμε στο λειτουργήμά και στο άτομό σας, επιτρέψατε μου δύο εκφράσεις μετά από τη δική σας παρέμβαση. Προσπαθήσατε να πνίξετε το θέμα ή να κάνετε ένα τεράστιο άλμα. Από τη μια πλευρά προσπαθήσατε να μας πείτε τα διάφορα κεφάλαια που θα είναι μέσα σε αυτό το πρόγραμμα δράσης, αλλά εμείς, και εγώ και οι συνάδελφοι, δεν μπορούμε παρά να χαρούμε που βρίσκουμε εκεί μέσα σε αυτόν τον κατάλογο τα βασικά από τις δικές μας προτάσεις. Μας δίνετε λοιπόν την απόδειξη ότι και μέσα στην Επιτροπή έχετε τα στοιχεία στη διάθεσή σας για να δημοσίευσε το πρόγραμμα δράσης σε όλες, με όλες τις συνιστώσεις. Όσο με αφορά λοιπόν, πιστεύω πως θα μπορούσαν να υπάρχουν οι εξή επεξηγήσεις. Για την πρώτη σας βράση στο δεύτερο τμήμα που λέει, αν κατάλαβα καλά τη μετάφραση, ότι δεν είναι ευνοϊκές οι συνθήκες. Πρώτη πιθανή συνθήκη είναι στο πλαίσιο της ΓΔ μεταφορών μια ανεπάρκεια τεχνικών πληροφοριών τα στοιχεία που μας έδωσε ο κύριος Μπαρό στην πλαίσιο του πράσινου βιβλίου μας άφησαν να πιστεύουμε πως αντιθέτως έχει υπερβολικά πολλές τεχνικές πληροφορίες διάθεσή της η Επιτροπή. Δεύτερη υπόθεση, λέτε ότι δεν είναι κατάλληλες οι συνθήκες. Γιατί κάποια κράτη-μέλη είναι αντίθετα. Ναι, αλλά κύριε Επίτροπε, από όσο γνωρίζω η Επιτροπή είναι ανεξάρτητη από τα κράτη-μέλη. Δεν μπορώ ούτε για μια στιγμή να πιστέψω ότι υποχαρίσατε στην πίεση ορισμένων κατορμελών. Μένει μια τρίτη υπόθεση γιατί ευνοϊκέ συνθήκε δεν πληρούνται. Μα είπατε ότι και ακόμα στο πλαίσιο τη Κομισιόν υπάρχουν ε, αποκλήσει που σα εμποδίζουν να μα υποβάλλετε αυτό το πρόγραμμα δράση. Ελπίζω για όνομα του Θεού, πω όχι. Και τέλο, θέλετε να αρνηθείτε τη συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να τον βάλετε για την επόμενη χρονιά, δεδομένων των εξαίρετων εκθέσεων που έχουν ε, τροφοδοτήσει τις σχέσεις μας με τον Αντιπρόεδρο Μπαρό κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το πράσινο βιβλίο, δεν τολμώ να το πιστέψω. Κύριε Πρόεδρε, λίγες εβδομάδες μας χωρίζουν από τις εκλογές. Αυτό το πρόγραμμα δράσης, κατά την άποψή μου, θεωρεί, ε, αποτελεί ένα εξέρδο παράδειγμα για να δείξουμε στους πολίτες μας πόσο η Ευρώπη, με σεβασμό στην επικουρικότητα, βρίσκεται κοντά στα προβλήματα υγείας τους, τα οποία σας επαριθμίσατε. Και λυπούμε βαθύτατα για αυτή την καθυστέρηση και ελπίζω, πως και οι συνάδελφοι, πώς θα μπορέσετε να διορθώσετε την κατάσταση όσο γίνεται πιο σύντομα. Σας ευχαριστώ. Πράσινη, ο κύριος Κράμερ, για 1,5 λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Η μόνιμη καθυστέρηση και η δική σας απάντηση δεν είναι αποδεκτή, Επίτροπε. Γιατί ο χρόνος πιέζει. Στο πλαίσιο των κλιματικών αλλαγών, οι αστικές μεταφορές αποτελούν μια πολύ μεγάλη συνιστώση, συνιστώση καθώς ευθύνονται για πάνω από το 50% των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Και μόνο με ευρωπαϊκή πολιτική θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο. Οι περισσότερες αστικές μεταφορές είναι λιγότερο από 6 χιλιόμετρα. Είναι πραγματικά αποστάσεις που θα επέτρεπαν να χρησιμοποιήσει κανείς το λεωφορείο, το τραμ, το τρένο ή να μετακινηθεί με τα πόδια. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει τα κράτη και τις πόλεις. Μας πρότειναν διάφορα κείμενα, πιο δεσμευτικά, το πράσινο βιβλίο ή την έκθεση ΡΑΚ. Όλα αυτά δεν έχουν πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Βλέπουμε ότι μέχρι στιγμής το 60% των ευρωπαϊκών κονδυλίων που αφιερώνονται στις μεταφορές αφιερώνονται στις οδικές μεταφορές. Μόνο το 40% στις δημόσιες μεταφορές και στο σιδηροδρόμους. Εμείς θέλουμε να αντιστρέψουμε την τάση όπως το ζήτησε και το Κοινοβούλιο για το πακέτο για τους σιδηροδρόμους. Εμείς θέλουμε μόνο να δοθούν επιδοτήσεις αν, υπάρχουν αν υπάρχει πρόγραμμα για βιώσιμη ανάπτυξη για τις αστικές μεταφορές και θέλουμε να περιορίσουμε την ταχύτητα ε, στα 30 χιλιόμετρα στις πόλεις και ορισμένες μόνο να έχουν μια ψηλότερη ταχύτητα. Καλό θα ήταν αυτό για το κλίμα και καλό θα ήταν επίσης για την αντιμετώπιση της νησιμότητας στους δρόμους. Ο κύριος Βλάσακ τώρα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι. Κρίμα που καθυστέρησε να δημοσιευθεί αυτό το έγγραφο, αλλά και το πρόγραμμα δράση. Γιατί, όπω είπαμε, όπω προαναφέρατε, έχουμε τόσου Ευρωπαίου συμπολίτες μας ζουν στι πόλει και οπότε ε, φυσικά και είναι πάρα πολύ σημαντικό το να του εξασφαλίσουμε τη, κάποιες μεταφορές, δημόσιες μεταφορές, οι οποίες όμως να είναι και φιλικές στο περιβάλλον. Οπότε, όταν γίνει η δημοσίευση του εγγράφου, ελπίζω ότι δεν θα περιγράφει μόνο κάποιες ε, τάσεις, και καταστάσει, αλλά να έχει και την αξιολόγηση της χρήσης ε, κάποιων μορφών μετακίνησης, όπως ε, τη μετακίνηση κάποιου πεζή ή με ποδήλατο και έτσι να μπορέσει ο καθένας να δει τι είναι το πιο κατάλληλο για κάθε πόλη, για κάθε δήμο, για κάθε κοινότητα και αυτή θα πρέπει να είναι η βασική μας προσέγγιση. θα πρέπει να ξεχωριστούν βέβαια κάποιοι πόροι τα ταμεία και έτσι να βοηθεί ε, αυτό το όραμα. Κυρία Τζοντίνη, δύο λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, εγώ Συμφωνώ πολύ με τα όσα είπαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι. Το αστικό περιβάλλον αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεύει ένα πολύ μεγάλο τμήμα της ζωής μας και όχι μόνο για αυτούς που ζουν ε, σε πόλεις μεγάλων ή μεσαίων διαστάσεων. Τα στοιχεία που δόθηκαν από την Επιτροπή στο Πράσινο Βιβλίο για μια νέα κουλτούρα στην αστική κινητικότητα δείχνει ότι το, ε, το 70% του ευρωπαϊκού πληθυσμού ζει στις πόλεις ε, και έχει μεγάλη συμβολή στο ΑΕΠ. Τους τελευταίους μήνες αυτά τα στοιχεία δεν έχουν αλλάξει και θα πρέπει ωστόσο να λάβουμε υπόψη πως τα προβλήματα συμφόρησης ε, κυκλοφορικής συμφόρησης στις μεγάλες πόλεις συνεχίζουν να αυξάνονται, όπως επίσης τα προβλήματα τα περιβαλλοντικά παραμένουν στην επικαιρότητα, όπως επίσης δεν είναι δυνατόν να ξεχάσουμε τις μεγάλες προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τελευταία για το πακέτο για το κλίμα. Υπάρχουν πολλαπλά στοιχεία. 2.000, 2 ε, δις ε, ευρώ δαπανήθηκαν για την περιφερειακή ανάπτυξη στην προηγούμενη θητεία και από το 2007 μέχρι το 2013 προβλέπονται 8 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υποστηρίξει αυτή την παρέμβαση. Θα πρέπει να είναι πραγματικά σημαντικό να υπάρχει μια κοινή πολιτική, ένα πρόγραμμα δράση σφαιρικό. Φυσικά με σεβασμό της επικουρικότητας και των αρμοδιοτήτων των ε, χωρών και των τοπικών αρχών. Τα ωφέλη που θα προκύψουν είναι προφανή και δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς ένα πρόγραμμα τέτοιο εύρους δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί. Προς αυτή την κατεύθυνση ε, προχωρούν ε, οι προφορικές ερωτήσεις που υποβλήθηκαν από την, τον πρόεδρο της Επιτροπής μεταφορών, την οποία υποστηρίζουμε και εμείς από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πιστεύω ότι πραγματικά η Επιτροπή θα θέλει να δώσει συνέχεια στη δημοσίευση του προγράμματος για την δράση για την αστική κινητικότητα με όλες τις θετικές συνέπειες που θα πέραν από αυτό. Ο κύριος Όλμπρεχτ για δύο λεπτά. Κυρίε και κύριοι, βεβαίω είναι αυτονόητο ότι ένα τέτοιο θέμα το οποίο αφορά τι δημόσιε μεταφορέ είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη, όσον αφορά το περιβάλλον. Επίση, ε, αυτό είναι αναμφίβολο και δεν θα πρέπει κανεί να ε, το αμφισβητεί τώρα. Όσον αφορά την πορεία την οποία κάναμε σε σχέση με την πράσινη βίβλο, ανέγυψαν και άλλα προβλήματα τα οποία τα ανέφεραν συνάδελφοι, κυρίως όσον αφορά την κατανομή των αρμοδιτήτων μεταξύ των ε, εθνικών αρχών, των τοπικών αρχών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και υπήρξαν κάποια ερωτήματα σε σχέση με το κατά πόσον θα πρέπει τέτοια θέματα τοπικής ε, υφής να τα ρυθμίζει η Ευρώπη ή θα πρέπει να τα αφήσει στις τοπικές ε, και εθνικές αρχές. Γιατί εγώ σας τονίζω ότι στη διάρκεια των εργασιών μας ανέκυψε το τι θα γίνει με κάποιες δραστηριότητες που θα εξωθήσουν τελικά τους δήμους, τις πόλεις να προχωρήσουν σε ανάληψη δράσης. Πώς θα βοηθήσουμε τέλος πάντων τις πόλεις και το ερώτημα επίσης είναι τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποιο είναι το σχέδιο το οποίο έχει για αυτό το ζήτημα. να αναλυφθεί η δράση δυναμική, να διερευνήσει πρώτα πρώτα τι πρεσβεύει ο κόσμος. Έδειξαν εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από την πρώτη τη αντίδραση που ήταν αρκετά συγκρατημένη. Προχώρησε και ακόμα όμως δεν έχει προκύψει σαφώς τι θα κάνει. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα λήψης κάποιων συγκεκριμένων αποφάσεων. Ελ έχετε δύο λεπτά κύριε. Σας ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι είμαι και εγώ αγνακτισμένος που και άλλοι συνάδελφοι σε σχέση με αυτό το οποίο είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίτροπε, φυσικά είναι αυτονόητο και είναι δικό σας καθήκον και αρμοδιότητά σας να, να αναλάβετε κάτι ε, κάποιες πρωτοβουλίε για αυτή την κινητικότητα. Όμως, εμείς θέλουμε κάτι παραπάνω, θέλουμε ένα λεπτομερές, ένα ενδελεχές πρόγραμμα δράσης. Εκεί να περιγράφονται κάποια μέτρα, κάποιες πολιτικές που προτίθεστε να ασκήσετε τα μέσα επόμενα χρόνια. Οπότε, κατά αυτόν τον τρόπο, να μπορέσετε να μας βοηθήσετε να ε, προβληματιστούμε και να δούμε ποιος και πόσο μπορεί να βοηθήσει από τους εμπλεκόμενους. Άρα από σας περιμένουμε να ε, μιλήσετε στους ανθρώπους της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι να κάνετε ε, για αυτό το πρόγραμμα δράσης. Ακούσατε σήμερα ε, πόσο πιέζει το θέμα, πόσο μας ενδιαφέρει. εκλογές έρχονται. In al και σαφώς επομένω προέκυψε ότι η κινητικότητα είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα που στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης. Όλοι έχουμε αυτό το πρόβλημα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης ε, μπορεί να διαρματίσει σημαντικό ρόλο όταν έρθει η ώρα τη ε, ανέβρεση κάποιων λύσεων για όλε αυτέ τι ευρωπαϊκέ πόλει. Θέλουμε κάποιε λύσει με βάση τι νέε τεχνολογίε. Θέλουμε ε, την καινούργια πρότυπα να διαδοθούν και επίση να διωθούν οι άριστε των πρακτικών. Οπότε μπορεί να βοηθήσει η Ένωση για τα νέα προγράμματα για τι μεταφορέ, μπορεί να βοηθήσει και απλώ βέβαια χρηματοδότηση. Οπότε, για άλλη μια φορά, παρακαλώ κύριε Επίτροπε, σα παρακαλώ πάρα πολύ, να ξανασκεφτείτε αυτό το οποίο μα είπατε. Εξασφαλίστε ότι θα υπάρξει ένα πρόγραμμα δράση βράδυ Κομισιόν όσο γίνεται ε, συντομότερα. Ευχαριστούμε κύριε Χαντράβη. Κυρία Τικάουτρο έχει το λόγο για το ΚΑΤΣΔΙ και έχετε το λόγο για ένα λεπτό Ευχαριστώ κύριε Επιτροπέ. Κύριε, κύριε Πρόεδρε, το πρόγραμμα δράση για την κοινότητα είναι αναγκαιότητα για τις πόλεις Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 70% των πολιτών αναμένουν μια εξέλιξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά. Ποια είναι η απάντηση της Κομισιόν Υπάρχει ένα έντονο κόστος που προβλέπεται από τη συμφόρηση. 1% του ΑΕΠ ελέγχθη ότι κοστίζει αυτό. Για να μειωθούν όμως οι συμφορέ αυτέ, θα πρέπει να υπάρχουν επενδύσεις σε αποτελεσματικά μέσα μαζικής μεταφοράς. Ε, η Πράγα είναι μια παραδειγματική πόλη. Έχουμε οικολογικά λεωφορεία για τις μεταφορές των ατόμων στα αστικά κέντρα. Εγώ ε, ζητώ να χρησιμοποιηθούν για τέτοια μέτρα και μέσα από τα διασωτικά ταμεία για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την κινητικότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλοι πρόεδρες. Κυρία Επίτροπος. Madam President, ε, Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις συμβουλές σας, συμβολές σας και θα μεταβιβάσω όλα όσα είπατε τον Αντιπρόεδρο κύριο Ταζάνη, ο οποίος ξέρω ότι εξακολουθεί να παραμένει δεσμευμένος αυτά. Το πρόγραμμα δράσης πραγματικά είναι στο πρόγραμμα εργασία τη Κομισιόν για το 2009 και εκείνο ο ίδιο προσωπικά έχει αναλάβει τη δέσμευση να προωθήσει το πρόγραμμα δράση αυτό. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτά που είπατε θα ληφθεί σοβαρά υπόψη από τον Αντιπρόεδρο κ. Τεζάνη. Ξέρω ότι έχει ολοκληρωθεί η μελέτη επιπτώσεων και όπως σας είπα το πρόγραμμα δράσης είναι στο πρόγραμμα εργασίας της Κομισιόν και θα το προωθήσουμε φέτος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρος. Κλείνει η συζήτηση. Σύμφωνα με την ημερησιακή περνάμε στην προφορική ερώτηση προς την Κομισό για την αναθεώρηση της ανακοίνωσης για τις ραδιοπλοκές μεταδόσεις, κρατικέ ενισχύσει για τη δημόσια υπηρεσία διαδρομικών αναμεταδόσεων. Και θέλω να δώσω το λόγο αμέσως στον συντάξοντα, τον κύριο Φίσερ, για 5 λεπτά.